Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα λοιπόν περνάμε στην ε, ψηφοφορία και επειδή έχουμε καθυστερήσει οι προφορικές επεξηγήσεις ε, δεν θα λάβουν χώρα αμέσως μετά την ψηφοφορία αλλά θα λάβουν χώρα μετά την τελική συζήτηση σήμερα το βράδυ. Και επίσης θέλω να ανακοινώσω ότι η επόμενη συζήτηση θα ξεκινήσει ευθύ αμέσως την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ψηφοφορία. Είναι η έκθεση Ντενανό και είναι ονομαστική ψηφοφορία. Μία και μόνο ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι χειροκροτείτε γιατί κάποιοι συνάδελφοι ήρθαν καθυστερημένα. Μπα περιπτώσει, κλείνει τώρα η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται η έκθεση. Και περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Ολτσκοφ. Πρόκειται για την απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα, επόμενη έκθεση ψηφίζουμε επίσης για την έκθεση της κυρίας Ουλφσκοφ. Είναι η απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Αποσχόλησης, ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Συνάδελφοι, κοιτάξτε, είναι ονομαστική η ψηφοφορία και έκλεισε, τώρα έκλεισε. Εγκρίθηκε και αυτή η έκθεση και περνάμε τώρα την έκθεση ε, των κυρίων Όμπριθ και Τόμας. Πρόκειται για την απόφαση ε, για την ε, τροποποίηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 14-20. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε και αυτή η έκθεση. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για την γενοκτονία έναντι των Αρμενίων. Ε, επτά ομάδες έχουν καταθέσει το ψήφισμα με διάφορες τροπολογίες. Τροπολογία υπερθμών 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές Επίσης απορρίπτεται. Η 4, τροπολογία υπαρτημών 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης απορρίπτεται. Τροπολογία υπαρτημών 5, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης απορρίπτεται. Μισό λεπτό. Η πρόεδρος λέει ότι οι συνάδελφοι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το αποτέλεσμα, αλλά εντάξει, αν θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία υπαριθμών 5. Ψηφίζουμε τώρα παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε επίσης. Ναι. Βλέπετε, επιβεβαιώθηκε η δική μου η άποψη. Η 6 τώρα, το πλογή υπέρ 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εδώ πραγματικά χρειαζόμαστε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για την τροπολογία υπερτιμών 6. Ψηφίζουμε τώρα παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και τώρα Ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ παρακαλώ. Κατά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα λοιπόν περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία. Πρόκειται για το ψήφισμα για τη Διεθνή ημέρα των Ρωμά και για την γενοκτονία των Ρωμά κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα ψήφισμα που κατέθηκε από διάφορες πολιτικές ομάδες. Έχουμε δύο τροπολογίες με ονομαστική ψηφοφορία και ξεκινάμε με την πρώτη τροπολογία, την υπαριθμών 2 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Και η τροπολογία υπαρτιμών 1, επίσης με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Γκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες και Συνεχίζουμε με τις ανακοινώσεις, θα τις κάνω στα γερμανικά. Και θα περιμένω μέχρι να βγουν οι συνάδελφοι από την αίθουσα που επιθυμούν να βγουν. Αν έχετε καλοσύνη να βγείτε γρήγορα.